Ladies and Καλησπέρα σας. Να σας υπενθυμίσω και να υπενθυμίσετε και στους συναδέλφους που θα έρθουν αργότερα ότι αργότερα θα ψηφίσουμε και όσοι δεν έχουν τις κάρτες τους μαζί τους παρακαλώ να βεβαιωθούν ότι μέχρι τη στιγμή που θα ψηφίσουμε πρέπει να τις έχουν προμηθευτεί. Το πρώτο θέμα είναι λοιπόν η ημερήσια διάταξη δεν έχετε αντιρρήσει υποθέτω γίνεται δεκτή. Στις ανακοινώσεις του Προέδρου τώρα να πω ότι παρέχεται διαμηνία σε όλες τις γλώσσες εκτός από γοηδελικά και κροατικά. Λοιπόν, σε σχέση τώρα με την υπηρεσία καινοτομίας η Γενική Διεύθυνση ITEC θέλει να κάνει κάποια πειράματα αυξημένης πραγματικότητας στη λήψη εικόνων. Και γι' αυτό ακριβώς θα υπάρξει ένα traveling 360 μοιρών. Νομίζω ότι θα το καταλάβατε αυτό. Ίσως για μένα θα ήταν καλύτερα να σταθούν περισσότερο στο πρόσωπό μου σε ευθεία, αλλά εν πάση περιπτώσει η διαδικασία αυτή δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει προβλήματα, αν υπάρξει κάτι θα επανέλθω. Έχουμε επίσης να πούμε για την ακρόση του King, υπευθύνου για θέματα ασφαλείας. Ξέρετε ότι έγινε πρόταση ο Σερ Τζούλιαν να είναι ο επόμενος Βρετανός Επίτροπος. Να σας πω ότι η ακρόαση για το Σερ Τζούλιαν θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Οι ακροάσεις αυτές θα ξεκινήσουν στις 7 και θα πάνε μέχρι τις 10. Μετά θα συναντηθούν οι συντονιστές το πρωί στις 13 για να αξιολογήσουν τις ακροάσεις και να μπορέσει ο πρόεδρος της Επιτροπής να ενημερώσει τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου για να υπάρξει απόφαση και της Ολομέλειας την ίδια εβδομάδα. Όλα αυτά γίνονται πολύ βιαστικά, αλλά ελπίζω όλοι να καταθέσετε τις ερωτήσεις που έχετε στο νου σας. Τώρα για τις συστάσεις των συντονιστών, ορισμός εισηγητών, Σαρτζεντίνη, η για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροπολογεί την οδηγία 215-849 για την αποφυγή χρήσης των κοινοτικών πιστώσεων για τρομοκρατικές ενέργειες και για άλλου είδους μορφές ε, κεφάλαιο επίσης για τους κανονισμούς σε σχέση με την δυνατότητα πολιτών τρίτων χωρών και, και στην περίπτωση επίσης αυτών οι οποίοι είναι άνευ τους απάτριδες, σχετικά με τη δυνατότητα απόκτησης διεθνούς, της ιδιότητας διεθνούς προστασίας. Ο κύριος Μωράες με την απλοποιημένη διαδικασία του άρθρου 50 είναι εισηγητής για τη Συμφωνία Στρατογική Συνεργασία ανάμεσα στους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Άμυνας της Κίνας και την Ευρωπόλ. Φεράρα επίσης και για την απόσυρση της οδηγίας 32-2013. Η κυρία Ιντβελτ έχει οριστεί επίσης συσυγήτρια για τις συνθήκες υποδοχής, τροπολόγηση της 33-2013 σχετικά με την υποδοχή αυτών που ζητούν να τύχουν διεθνούς προστασίας. Έχουμε επίσης συσυγητές για γνωμοδοτήσεις, η κυρία για τον συντονισμό ορισμένων ρυθμίσεων ή διοικητικών πράξεων σε διάφορα κράτη-μέλη για την παροχή υπηρεσιών ε, του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Η, κυρίου η κυρία μάλλον Παγκαζαρωτώντα για την προστασία αυτών οι οποίοι καταδίδουν προς το δημόσιο συμφέρον ε, εμπιστευτικές πληροφορίες. Ζητώ από την Επιτροπή να δεχθούν τους συστάσεις αυτές σύμφωνα με το άρθρο 205 της 6ης Ιουνίου 2016. Σας είπα να πάρετε τις κάρτες σας γιατί θα γίνει ψηφοφορία αργότερα στις 5.30. Αλλά θα επανέλθουμε για τα θέματα αυτά σε έφετο χρόνο. Περνάω λοιπόν στο σημείο 3. Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα των ποινικών, Eurojust θα γίνει μια παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για το 2015 από την κυρία Κόνιγκς, πρόεδρο του Eurojust. Η παρουσίαση της κυρίας Κόνιγκς θα ακολουθηθεί από ανταλλαγή απόψεων. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Ε, νιώθω ιδιαίτερη τιμή με την ευκαιρία που μου δίνεται να σα παρουσιάσω την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τη Eurojust για τι δραστηριότητε του 2015. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω πάνω από του 350 υπαλλήλου τη Eurojust ε, που εργάστηκαν αργοδό πέρυσι για να, να δώσουν τη μάχη αποτελεσματικά κατά της ε, τρομοκρατίας, χρηματοδότησης τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος και σε όλα αυτά τα θέματα της ε, ποινικής συνεργασίας. Νομίζω ότι μετά τις τερινές διακοπές μπορούμε να πάρουμε μια νέα φόρα και να ε, ενισχύσουμε τις ε, αντιδράσεις μας αυτές τις απειλές που αντιμετωπίζουμε και στην ασφάλεια και από το οργανωμένο έγκλημα. Είναι καλή ώρα για έναν απολογισμό, να δούμε πού βρισκόμαστε και προς τα πού βαδίζουμε. Ευχαριστώ θερμά όλους όσους στήριξαν τη Eurojust στην αποστολή της. Βλέπουμε εδώ από τη διαφάνεια τα στοιχεία που μιλούν από μόνα τους. Το 2015 είχαμε μια αύξηση κατά 23%, πάνω από 23% των υποθέσεων που έφτασαν στην Eurojust στη σχέση με πέρυσι, το 2014, πρόπερσι μάλλον. Το 2015 ασχοληθήκαμε με 2.214 υποθέσεις. Φαίνεται δηλαδή ότι η Eurojust και οι υπηρεσίες της παρέχουν πολύ χρήσιμες υπηρεσίες, κάτι που αναγνωρίζετε και η μόνη ανησυχία που έχουμε αφορά την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων μετά την αύξηση των, του των εργασιών. Γιατί αυτή η αυξητική πορεία του των εργασίας θα συνεχιστεί και το 2016. Δεν φανταζόμαστε να μειωθούν οι εγκληματικέ δραστηριότητες ε, το, του επόμενου μήνε ή χρόνια. Μάλλον το αντίθετο. Οπότε με τους ίδιους πόρους έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ περισσότερε υποθέσει. Εδώ βλέπετε και άλλα στοιχεία. Όπως σας είπα, ε, επεξεργαστήκαμε πάνω από 2.200 υποθέσεις. Η ανάμειξη των τρίτων χωρών μελών επίσης ήταν σημαντική. Είχαμε περίπου 298 υποθέσεις με ανάμειξη τρίτων χωρών στις βασικές δραστηριότητες ε, ε, δικαστικού συντονισμού και δικαστικής συνεργασίας και αναφίβολα, κάτι που φαίνεται και από τα στοιχεία, έχουμε τρεις βασικές κατηγορίες εγκλήματος ε, την τρομοκρατία, την λαθροδιακίνηση, το έγκλημα στο κυβερνοχώρο, αλλά και την εμπορία ανθρώπων, απάτη, διαφθορά και κινητές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό αντιμετωπίζουμε κυρίως και φαίνεται και από τα στοιχεία και άλλων οργανισμών. Και αυτό δείχνει και ο αριθμός των υποθέσεων ε, με την αντίστοιχη εμφάνιση των διαφόρων αυτών φαινομένων κλιματικότητας. Εμείς οργανώνουμε και συντονιστικές ε, συναντήσεις. Είχαμε πάνω από 274 τέτοιες ε, συντονιστικές συνεδριάσεις και αν συνδυάσουμε αυτό το στοιχείο με τα περσινά στοιχεία, διαπιστώνουμε ότι η αύξηση ήταν γύρω στο 40%, 39% για την ακρίβεια αύξηση στον αριθμό των συντονιστικών συνεδριάσεων. Κάτι που σημαίνει όλο και περισσότεροι αστυνομικοί, ανακριτέ, ε, εισαγγελεί και δικαστέ είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε τέτοιε συντονιστικέ συνεδριάσει και να εξετάζουν από κοινού με άλλου συναδέλφου ε, τα φαινόμενα αυτά τη εγκληματικότητα. και βλέπουν την προστιθέμενη αξία αυτού του συντονισμού. Θα πρέπει λοιπόν να, δρούμε και να αντιδρούμε εγκαίρω. Και μάλιστα στις συντονιστικές συνεδριάσεις φαίνεται ότι χρειάζεται η θέσπιση στρατηγικών και η αποστολή και στοιχείων προς τα συντονιστικά κέντρα. Δείχνει αυτή την άμεση αντίδραση που έχουμε. Και μάλιστα το 2015 οργανώσαμε 13 τέτοια συντονιστικά κέντρα. Και μία από τις ένα από τα βασικά μας συντονιστικά κέντρα είναι αυτό που αφορά την, την τρομοκρατία και μάλιστα στήθηκε ε, μία μέρα πριν την τρομοριστική επίθεση στο Παρίσι και αποτρέψαμε περαιτέρω ε, τέτοιες απειλές μόνο και με ε, συντονισμό μεταξύ των δικαστικών και αστυνομικών αρχών. Επίσης, είχαμε πάνω από 100 τέτοιες κοινέ ερευνητικές ομάδες, ΑΤΖΙΤ, και χρηματοοικονομική υποστήριξη σε 68 τέτοιες κοινέ ομάδες έρευνας. 68 τέτοιες τις στηρίξαμε οικονομικά, γιατί οι κοινέ ε, ερευνητικέ ομάδες είναι η Rolls Royce της αμοιβέ ε, δικαστικής αρρωγής. Και είναι η ατμομηχανή αυτή τη προσπάθεια που κάνουμε για την εφαρμογή του κράτους δικαίου. Επίσης, ε, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ε, είναι πολύ επιτυχημένο. Είχαμε 292 τέτοιε περιπτώσεις και συμβάλαμε στην εκτέλεση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης. Και μάλιστα ο προπολογισμό μέχρι το 2015 ήταν 33.818.000. Ακούγεται ω υψηλό ποσό, αλλά πραγματικά δεν είναι, γιατί εκτελέστηκε σχεδόν πλήρω Το ποσοστό εκτέλεσης ήταν 99,86% για το 2015. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια και βλέπουμε με μεγεθυντικό φακό το έγκλημα και διαπιστώνουμε ότι αυτό που προσφέρουμε είναι αυτό που χρειάζονται οι δικαστικές αρχές των κρατών μελών. Γιατί προσφέρουμε υπηρεσίες, στήριξη, ε, συμβάλλουμε στη θέση στρατηγικών, ε, επιταχύνουμε την, εκτέλεση, την εφαρμογή της δικαστικής συνδρομής και μάλιστα έχουμε επαφές και με τρίτες χώρες που δεν είναι τόσο εύκολες οι επαφές. Και μόνο όταν έχουμε σωστέ επαφές με τους κατάλληλους ανθρώπους και σε τρίτες χώρες ε, έχουμε αποτελεσματική συνεργασία. Ε, Δυτικά Βαλκάνια, Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή. Με τις χώρες αυτές ε, δημιουργούμε όλο και πιο έμπιστες επαφές Επίσης, εξαρτώμαστε από τις αιτήσει που υποβάλλουν οι δικαστικές αρχές των διαφερομένων κρατών μελών. Και είναι κοινά τα προβλήματα, τρομοκρατία, λαθροδιακίνηση, λαθρεμπόριο, έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Είναι κοινέ οι απειλέ και μάλιστα η έκταση των φαινομένων αυτών ε, είναι άνευ προηγουμένου και τα κράτη-μέλη έχουν κατακλειστεί από την προσπάθεια να ανταποκριθούν στο προσφυγικό φαινόμενο, αλλά και στην δραστηριότητε των αθροδιακινητών. Όλα τα κράτη-μέλη επίση αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των ξένων μαχητών. Αλλά και το ψηφιακό τομείο, το οποίο εκτελήσεται με τόσο ραγδαίους ρυθμούς που εξορισμού ε, όλα αυτά τα εγκλήματα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Οπότε πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, αυτές αποδείξεις και τεκμήρια. Έχουμε προβλήματα δικαιοδοσίας επίσης, σύγκρουση δικαιοδοσιών και αρμοδιοτήτων, κάτι που είναι το καθήκον των δικαστικών αρχών. Επίσης παρακολουθούμε και το σχέδιο δράσης για την ασφάλεια και για το, τη ε, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με τις προτεραιότητες ε, τα παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μάλιστα αναφέρουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στην έκθεση του 2015 και εμείς επικεντρωνόμαστε στις βασικές ε, προτεραιότητες που είναι έγκλημα στον κυβερνοχώρο, τρομοκρατία και λαθροδιακίνηση των μεταναστών. Φυσικά και το ξέπλυμα χρήματος είναι πολύ σημαντικό και πολύ και η διαφθορά, το περιβαλλοντικό έγκλημα δεν μπορούμε να, αντιμετωπίσουμε, να παραμελήσουμε και αυτές τις μορφές εγκληματικότητας. Βέβαια έχουν είτε άμεση είτε άμεση σχέση και με τις προηγούμενες προτεραιότητες του οργανωμένου εγκλήματος και αυτό το διαπιστώνουμε καθημερινά. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Εμείς ε, το 2015 συνεχίζουμε για τρίτη συνεχή χρονιά να επικεντρωνόμαστε στο φαινόμενο των ξένων μαχητών. Και μάλιστα συμμετείχαμε και στην παρακολούθηση των ε, ε, ε τρομοκρατικών επιθέσεων και στο Παρίσι και στη Δινησία. Και φυσικά από την αρχή συμμετείχαμε στην παρακολούθηση αυτών των επιθέσεων και συνεχίσαμε και την ανάμειξή μας και στη συνέχεια στις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες και σε άλλες τέτοιες. Είχαμε και ένα άτυπο δίκτυο ε, εισαγγελέων αντιτρομοκρατίας. Είναι ένα άτυπο δίκτυο αυτό των εισαγγελέων αντιτρομοκρατίας και συναντιόμαστε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές, βέλτιστες πρακτικές, αντλούμε διδάγματα από τις εμπειρίες μας. Επίσης έχουμε και το monitor για τις καταδικαστικές αποφάσεις σε θέματα τρομοκρατίας και βλέπουμε τις πιο εμβληματικές τέτοιες καταδίκες ε, στην τρομοκρατία. Ε, προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις αδυναμίες, ε, να επιταχύνουμε τα, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στις ποινικέ δίκες. Και αυτό το είδαμε και σε κάποιες υποθέσεις για τη Συρία. Επίσης, έχουμε και την εποπτεία, τη δικαστική εποπτεία για την πειρατεία στη θάλασσα. Μειώνεται αυτό το φαινόμενο, πολύ θετικό. Και μάλιστα αυτά που αρχικά είχαμε στις ανατολικές αφρικανικές ακτές έχουμε μεταβεί προς τις δυτικές αφρικανικές ακτές, αλλά με χαμηλότερη συχνότητα. Αλλά άλλες μορφές τρομοκρατίας δυστυχώς αυξάνονται. Τώρα, το εγχειρίδιο για τις χημικές, βιολογικές, ραδιολογικέ πυρηνικέ και απειλές στον κυβερνοχώρο έχει ετοιμαστεί. Είναι σημαντικές αυτές οι απειλές, CBRNE, γιατί είναι μια πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδου απειλέ χημικού, βιολογικού, ραδιολογικού, πυρηνικού ή ηλεκτρονικού χαρακτήρα από τρομοκράτε. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ αυτή την κατάσταση. Επίσης, πέρυσι είχαμε ε, συνάντηση με τους υπουργού Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και παρουσιάσαμε τα βασικά μας πορίσματα και τις ε, βασικά μας συμπεράσματα για πώς θα καταπολεμηθεί το φαινόμενο της ε, λαθροδιακίνησης μεταναστών. Επίσης, ε, με τους εισαγγελείς αντιτρομοκρατίας συζητήσαμε πέρυσι κάποια σημαντικά θέματα κατά πολέμηση της και η έκθεση από την ε, συνάντηση αυτή θα δημοσιευθεί τον Νοέμβριο και η παρουσίαση θα γίνει αργότερα. Συνεχίζουμε λοιπόν το έργο μας. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και οι πυλές είναι σοβαρότατες και ουσιαστικές. Οπότε δεν μπορούμε να σταματήσουμε την επαγρύπνηση ή τη συνεχή προσπάθεια καταπολέμησης αυτών των μορφών εγκλήματος και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι πολύ σημαντικό. Το 2015 ξεκινήσαμε μια υψηλή ε, εμβέλεια ε, συνάντηση συντονιστών ε, ειδικευμένων στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Έχουμε και το EC3, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εγκλήμα, για Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο. Και έχουμε και 8 εθνικά τέτοια σημεία επαφής που συμμετέχουν την ανάλυση των απειλών που αντιμετωπίζουμε σε νομικό και δικαστικό επίπεδο. Επίσης, έχουμε επαφές και με τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, για τα θέματα αυτά και μάλιστα ε, θα έχουμε τη συνεργασία με τον ειδικό επισταλμένο από τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, εισαγγελέα γιατί πολλά απορίσματα συγκεντρώθηκαν εκεί, θα μας βοηθήσουν έτσι σε άμεση αντίδραση Μάλιστα θα έχουμε και άλλη συνάντηση ειδικευμένων εισαγγελέων και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό δίκτυο τέτοιων ειδικευμένων ε, εισαγγελέων για το οργανωμένο έγκλημα με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να συστήσουμε αυτό το δίκτυο. Και είναι σημαντική αυτή η στήριξη από την Επιτροπή και η στήριξη που θα προσφέρει η Eurojust στη συνέχεια. Θέλουμε να γίνουμε γέφυρα με, με τις 28 ε, εθνικές δικαστικές αρχές που αντιμετωπίζουν ε, αυτό το περίπλοκο φαινόμενο των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Τώρα, για τη λαθροδιακίνηση μεταναστών. Έχουμε πολλά προβλήματα, όχι μόνο στα κέντρα καταγραφής, στα hot spots, όχι μόνο στις χώρες διέλευσης, ε, ούτε μόνο στις χώρες προορισμού. Σε όλες τις χώρες αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Ακούσατε τι έγινε στις, τον Αύγουστο του 2015 με ένα φορτηγό ψυγείο που βρέθηκε στην Αυστρία με 71 νεκρούς πια μετανάστες και το Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε ε, συντονιστική προσπάθεια με την Αυστρία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Γερμανία τις τέσσερις χώρες από τις οποίες διήλθε αυτό το φορτηγό ψυγείο, γιατί από την Αυστρία ξεκίνησε, ο, φο, οι φορτηγατζίδες ήταν βουλγαρικής καταγωγής, ο εγκέφαλος ήταν από την Ουγγαρία και ο προορισμός η Δυτική Γερμανία. Είδαμε ότι αυτό ήταν το τελευταίο ταξίδι το οποίο είχε προβλεφθεί με ανθρώπινα όντα. Στη σειρά βέβαια είχαν προηγηθεί άλλα τρία-τέσσερα. Και δυστυχώς συνέβη αυτό το οποίο συνέβη τον Αύγουστο του 2015 στην Αυστρία. Βέβαια ήταν εξαιρετικά περίπλοκη η κατάσταση. Είχαν ήδη ξεκινήσει αμέσως μετά τα πρώτα ταξίδια αυτής της οργάνωσης, τις πρώτες δραστηριότητες αυτής της οργάνωσης σε διάφορες χώρες και ο συντονισμός είναι κάτι το πάρα πολύ περίπλοκο, στο οποίο όμως έχουμε προχωρήσει αρκετά. Εμείς προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε και σε τακτικό επίπεδο και σε επίπεδο στρατηγικό. Έχουμε επίσης συνεργασία με συναδέλφους στα διάφορα hot spots, έχουμε συνεργασία με Έλληνες, με Ιταλούς συνεργάτες. Προσπαθούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα και να το εξετάσουμε και στρατηγικά, όχι μόνο σε απτό πρακτικό επίπεδο, Προσπαθούμε να δούμε αν πρόκειται για το οργανωμένο έγκλημα το οποίο διαμορφώνει αυτές τις διαδικασίες. Συγκρίνουμε τις ποινές ε, για τέτοιου είδους ενέργειες στις διάφορες χώρες. Τι συμπεράσματα βγάζει κανείς από τη σύγκριση αυτή, τι βήματα χρειάζεται να γίνουν έτσι ώστε να υπάρξουν πιο συγκεκριμένες αποδείξεις ε, για τις απαράδεκτες αυτές δραστηριότητες. Επίσης και στα πλαίσια του trafficking συνεχίζουμε να συναντώμεθα με εξειδικευμένους εισαγγελείς αναχώρα και έχουμε κυκλοφορήσει ε, την ε, έκθεσή μας ήδη ακριβώς για τα θέματα του trafficking. Ήδη από το 2015 Είχαμε 39 σημεία επαφής τα οποία είναι μοιρασμένα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε φτάσει το 16 σε 40, συνεργαζόμεθα πλέον και με την χώρα του Μεξικού. Συνεπώς λοιπόν ε, επικοινωνούμε με σωστό τρόπο με τις αρμόδιες αρχές και με ε, τη μεγαλύτερη δυνατή εμπιστευτικότητα. Έχουμε υπογράψει όπως γνωρίζετε και συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης με το Μαυροβούνιο και την Ουκρανία. Και περιμένουμε να τεθούν οι συμφωνίες αυτές σε ισχύ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζουμε τις προσπάθειες συνεργασίας και με άλλες χώρες. Ε, βασικές στιγμές ε, το 2016 είτε ότι καλωσορίσαμε τους Ελβετούς συναδέλφους που αποφασίστηκε το 2015 να συνεργαστούν στα πλαίσια της Eurojust μαζί με τους Νορβηγούς και τους Αμερικανούς νομίζω προσφέρουν πάρα πολλά στην λειτουργία της Eurojust. Βλέπετε τον αριθμό των περιπτώσεων με τις οποίες καλούμεθα να ασχοληθούμε, ο οποίος αυξάνεται συνεχώς. Τα θέματα της τρομοκρατίας, σαν παράδειγμα, αναφέρθηκα λίγο πριν. Σας είπα ότι μία μέρα πριν από την επίθεση στο Παρίσι είχαμε μία συνάντηση συνεργαστήκαμε με Ελβετούς, συνεργαστήκαμε με Νορβηγούς και το κάνουμε αυτό έτσι και αλλιώς και σε άλλο επίπεδο από το 2011 και καταφέραμε χάρη στη συνεργασία με όλους αυτούς και τους Νορβηγούς να συλλάβουμε 10 επιπλέον άτομα τα οποία κατηγορούνται για τρομοκρατικές ενέργειες διαφόρων ειδών. Και αυτή η προσπάθεια θα αποδώσει ακόμα περισσότερο. Και τέλος προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν σε οργανωτικό επίπεδο. Έχουμε συνεργαστεί όπως είπα και σε επίπεδο δημιουργίας περαιτέρω σημείων επαφής, contact points. Ε, μας επιβεβαίωσε το Συμβούλιο ότι οι προτεραιότητες τις οποίες θα έχουμε είναι πραγματικές προτεραιότητες, συμφωνεί με αυτές. Οι στόχοι τους οποίους έχουμε, προσπαθούμε να επιδιώξουμε την ολοκλήρωσή τους και σε επίπεδο Eurojust και σε επίπεδο των υπολείπων ευρωπαϊκών δομών. Εμείς περιμένουμε να γίνουν κινήσεις για την πλήρη ενσωμάτωση των ρυθμίσεων οι οποίες διέπουν τη Eurojust Φυσικά υπάρχει και ο κανονισμός για την Europol που είναι, ε, καλύπτει ένα χώρο με τον οποίο και εμείς ε, καλύπτουμε. Καλούμεθα να συνεργαστούμε πλήρως ε, και με την Europol και σε όλους τους τομείς και σε σχέση με, το, με τις λεγόμενες ποινικέ δραστηριότητες PIF, PIF. Και ταυτόχρονα συνεχίζουμε τις ε, προσπάθειες συνεργασίας και με τις τοπικές αρχές. Η πολιετής μας στρατηγική έχει τρεις βασικούς στόχους. Καταρχές λειτουργική ε, ε, ευρυθμία, οργανωτικές εξελίξεις, κάλυψη δηλαδή των νέων οργανωτικών αλλαγών Έχουμε κάνει κάποια βήματα, απαιτείται όμως να κάνουμε περισσότερα συνδυάζοντας με καλύτερο τρόπο τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Υπάρχει επίσης και μια κάποια δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουμε στον τομέα της συμβατότητας διαφορετικών διαδικασιών που ακολουθούνται στις διάφορες χώρες για τη συλλογή στοιχείων, την σύγκριση των στοιχείων αυτών και την χρήση τους. Και τέλος θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι, αποδοτικοί και ε, να βλέπουμε ακριβώς εμείς πού υπάρχουν θέματα ποινικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τους εισαγγελείς των διαφόρων χωρών. Το πρώτο εξάμεινο του 17 και αυτό είναι καλό, θα μετακομίσουμε γιατί τώρα είμαστε στριμωγμένοι σε δύο μικρά κτίρια κάτω από συνθήκες ασφαλείας περιθωριακά ικανοποιητικές. Νομίζω ότι τα πράγματα εξελίσσονται καλά. Έχουμε βέβαια κάποια θέματα είναι η κατάσταση δύσκολη σε σχέση με τους ανθρώπινους πόρους. Μας ζητάνε συνεχώς να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερο κόσμο, με μικρότερο ανθρώπινο δυναμικό. Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει την δυνατότητα αυτή και είδαμε ότι ε, πολλές εξωτερικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τύχει υποστήριξης από τα υπόλοιπα όργανα Είμαστε ένα ζωτικός μικρός κρίκος της αλυσίδας ε, που διασφαλίζει ε, θα έλεγα την ε, δυνατότητα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν μπορέσουμε να μεγενθύνουμε αν θέλετε και το ανθρώπινο δυναμικό μας φοβάμαι ότι ποτέ δεν θα είμαστε στο ύψος των απαιτήσεων και δεν θα επηρεάσουμε όσο μπορούμε τον τομέα της ασφάλειας. Στον τομέα της δικαιοσύνης βλέπουμε ότι οι αριθμοί αυξάνονται σταδιακά. Προβλέπετε, στην αρχή ήταν πάρα πολύ χαμηλή η αριθμή αυτή σε σχέση με ε, το ανθρώπινο δυναμικό που είχαμε στη διάθεσή μας έχουν πολλαπλασιαστεί χωρίς ιδιαίτερη αύξηση του προσωπικού σήμερα. Κανονικά θα πρέπει να αρχίσω να κλαίω σαν καλή νοικοκυρά και μάνα και να λέω ότι δεν μπορώ πια κάνουμε ό,τι μπορούμε αλλά παίζουμε πια ε, εις βάρος της ασφάλειας και είναι πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με όλα αυτά τα θέματα και τους στηρίζω. Βέβαια έχουμε καλύτερες μορφές στήριξης από τις εθνικές υπηρεσίες από το 2017 και μετά. Εμείς ζητάμε 3 εκατομμύρια επιπλέον, όχι για να μπορέσουμε να ξοδέψουμε περισσότερο, αλλά για να μετακομίσουμε. Γιατί θα πρέπει τους επόμενους 6 μήνες να καλύψουμε έξοδα ασφαλείας σε τρία κτίρια γιατί ο κόσμος θα μετακινηθεί από το ένα κτίριο στο άλλο από τον Απρίλιο και μετά, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχουν και επικοινωνίες οι οποίες να είναι απολύτως ασφαλείς και μη προσβάσιμες. Λοιπόν, συνεργαζόμαστε σε πάρα πολλούς τομείς με τη Europol, όχι μόνο στον τοπινικό τομέα, αλλά και γενικότερα σε θέματα τρομοκρατίας, Γι' αυτό λοιπόν προσπαθώ να το κάνω με κάπως ευγενικό τρόπο, αλλά θα ήθελα να, είμαι, ε, να δώσω περισσότερο δράμα σε αυτό το οποίο ζητάω. Θέλουμε την υποστήριξή σας γιατί απαιτείται να κάνουμε περισσότερα. Ευχαριστώ. Πολύ περιεκτική παρουσίασή σας. Θα, θα ακολουθήσει η συζήτηση. Είπατε storm in a glass of water. Storm με τι λέμε στα αγγλικά, γιατί εμεί πίνουμε τσάι, οπότε βλέπουμε τι καταιγίδε περισσότερο σε φλιτζάνι τσαγιού και όχι σε ποτήρι. Πάντω καταλάβαμε τι εννοούσατε. Ποιο θα ήθελε πρώτα στο λόγο, παρακαλώ, παρατηρήσει σχόλια μετά την παρουσίαση τη αιτήσια έκθεση Eurojust. Κύριε Κρίσπεκ. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Διευθύντρια για αυτή την παρουσίαση ταχύτατη η οποία στηρίζει το πολύ λεπτομερές έγγραφο που μας έστειλε για την της ε, έκθεση του 2015. Φυσικά όλοι στηρίζουμε την ε, αύξηση των υποθέσεων που αντιμετωπίζει η Eurojust και καταλαβαίνουμε και την έκκλησή σας για στήριξη αλλά και για την ε, χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων ε, της ε, υπηρεσίας της Eurojust από όλους μας. Όλοι είμαστε πεπισμένοι ότι πρόκειται για κάτι το καθοριστικό σε σχέση με αυτά που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη και η Ευρώπη γενικότερα και φυσικά πρόκειται και για μια πραγματική απάντηση συντονισμένη σε σχέση με αυτά τα δραματικά γεγονότα που αντιμετωπίζουμε και ζούμε σε πολλά κράτη-μέλη, κυρίως ε, όμως σε κάποια από αυτά όπως στη χώρα μου, τη Γαλλία. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω. Αναφέρομαι στα συμπερασματικά σας σχόλια που αφορούν το δημοσιονομικό κομμάτι, τα μέσα που διαθέτεται και πριν από λίγες μέρες μας στείλατε αυτή την έκθεση και τις ανησυχίες σας. Πριν από λίγες μέρες η Επιτροπή μας, ασχολούμενη με θέματα προϋπολογισμού, στήριξε με μεγάλη πλειοψηφία, μέσω μιας τροπολογίας, την στήριξη αυτού του αιτήματό σας και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα σας αφήσουμε μόνους σας. Η Επιτροπή Προϋπολογισμού θα στηρίξει την τροπολογία αυτή το λέω αυτό για να σας πω ότι πραγματικά έχουμε ακούσει όλα αυτά τα αιτήματα που μας στείλατε με την επιστολή σας. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Για όλους τους Ευρωπαίους σήμερα το θέμα της ασφάλειας είναι καθοριστικό και είναι ακριβώς αυτό που κάνετε εσείς. Και βεβαίως για να υπάρξει ασφάλεια χρειάζεται ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν υπάρχει ούτε μία συνάντηση, ούτε ένα έγγραφο που να μην επαναλαμβάνει αυτή την προτεραιότητα, κάτι που πολλές φορές δεν ε, προωθείται όπως θα έπρεπε και το γαλλικό γραφείο της Eurojust μας ενημέρωνε πριν από δύο χρόνια, θυμάμαι, ότι ο αριθμός των στοιχείων που μεταβιβάζονται από τα 36 δικαστήρια με τα οποία επικοινωνεί η Eurojust στη Γαλλία είναι ελάχιστα. Μόνο ένα από αυτά τα 36 ανταλλάσσει πληροφορίες και στέλνει στοιχεία στην Eurojust. Δεν ξέρω αν η κατάσταση είναι παρόμοια και σε άλλα κράτη-μέλη και αυτή είναι και η ερώτησή μου. Άλλαξαν λίγο τα πράγματα από τότε. Η Γαλλία βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με πριν από δύο χρόνια υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών που βρίσκεται ουσιαστικά στην καρδιά της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Έχει λυθεί το θέμα αυτό, έχει εξελιχθεί η κατάσταση, υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σήμερα. Δεύτερη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω, πάντα στο θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών, γιατί βεβαίως επαναλαμβάνω ότι είναι κάτι που απασχολεί όλους τους Ευρωπαίους και όχι μόνο τα θεσμικά όργανα. Υπάρχει καλή βέλτιστη ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχει πρόσβαση των κρατών μελών μέσω του συστήματος ε, CMS στις ε, πληροφορίες Eurojust. Ξέρω ότι πάνω από τα μισά κράτη-μέλη δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο αυτό και τις πληροφορίες αυτές. Κάνω λάθος, είναι σωστές οι πληροφορίες μου ή έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Τελευταία ερώτηση που απαντήσατε εν μέρη στην παρουσίασή σας είναι το θέμα της συνεργασίας με τα τρίτα, με τις τρίτες χώρες. Μιλήσατε για 40 χώρες στον κόσμο. Είναι κάτι το απαραίτητο, το σημαντικό και το πολύ επίκαιρο. Στην τελευταία συνάντηση που είχαμε μαζί σας μιλήσαμε και για τις συμφωνίες συνεργασίας που είχαν υιοθετηθεί το 2016 και στην έκθεση δραστηριοτήτων σας είχατε αναφερθεί στην Αλβανία, στη Σερβία, στην Τουρκία, το Ισραήλ, τη Βραζιλία, Κολομβία, Μεξικό, Γεωργία, ολοκληρώνω πρόεδρε, για προτεραιότητες όσον αφορά τη συνεργασία και η ερώτησή μου είναι αν με αυτές τις τρίτες χώρες έχουν προσχωρήσει οι συμφωνίες συνεργασίας γιατί θεωρώ ότι όσον αφορά τη Σερβία και την Αλβανία είναι προτεραιότητες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Πρόεδρε του Eurojust για την παρουσίαση. Είναι πολύ σημαντική πλατφόρμα συνεργασίας η Eurodust μεταξύ των ε, αστυνομικών ε, και δικαστικών αρχών των κρατών μελών. Και ε, είδαμε ότι έχετε δημοσιονομικά προβλήματα με μικρό προϋπολογισμό για να αντιμετωπίσετε ένα ευρύ φάσμα μορφών εγκλήματος. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γνώμη έχετε για τον κανονισμό που έχει εγκριθεί και δεσμεύει τα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της εμπορίας ανθρώπων. Επίσης, η Eurojust έχει κάνει τη δική της αξιολόγηση του κανονισμού για την ποινική δικονομία. Δηλαδή, υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό αποτελεσματικότητας. Υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ Βελγίου και Γαλλίας μετά τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις των Βρυξελών και πολλοί άσκησαν κριτική για τον τρόπο που ασκείται το δίκαιο και η δικαστική πρακτική στο Βέλγιο απέναντι σε τόσο επικίνδυνες μορφές ε, εγκλήματος όπως είναι η τρομοκρατία. Ερωτώ λοιπόν εσείς ε, προσωπικά και η Eurojust ως θεσμικό όργανο έχει κάνει τη δική της ανάλυση για την ε, ποινική δικονομία και το πώς ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η εγκληματικότητα. Επίσης, πώς εκτιμάτε τον κανονισμό σε ό,τι αφορά το ποινικό, τις ποινικές ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της εμπορίας ανθρώπων. Γιατί Πιστεύετε ότι θα γίνουν κάποιες διορθώσεις στο θέμα της αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων. Και πιστεύετε ότι η νέα οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα υποδιάσει με καλύτερα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε στην Ευρώπη πιο αποτελεσματικά το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ κύριε Γκόμες. Σας ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε και ευχαριστώ πολύ για την πολύ ε, λεπτομερή σας παρουσίαση της ε, ετήσιας έκθεσης της Eurojust. Εδώ όμως αναφερόμαστε στο 2015. Ήδη έχει προχωρήσει όμως το 2016. Και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία της συνάντησής μας για να αναφερθώ στις συστάσεις για το μέλλον και στα συμπεράσματά σας. Τι συμβαίνει δηλαδή ήδη ενώ βρισκόμαστε στο 2016. Και θα ήθελα να σας ε, κάνω μια ερώτηση. Μιλήσατε για τα εγκλήματα, για την εμπορία ανθρώπων, ε, την ε, λαθροδιακίνηση και την παράνομη μετανάστευση. Τι συστάσεις κάνετε στα κράτη-μέλη, σε εμά εδώ, δια... δι θεωρείται ότι επειδή δεν υπάρχουν νόμιμες οδοί μετανάστευσης και κυκλοφορίας υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δεν έχουν δηλαδή εναλλακτικέ λύσεις αυτοί οι άνθρωποι από το να αφήσουν τις τύχες τους, τις ζωές τους στους διακινητές. Και τελικά δίνουμε δουλειά σε αυτούς τους ε, λαθροδιακινητές με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα να ακούσω την απάντησή σας. Επίσης, όσον αφορά την νόμιμη λαθροδιακίνηση, όσον αφορά αυτές τις νομιμοποιήσεις παράνομων ε, πόρων με όλα αυτά τα προγράμματα. Ξέρω ότι υπάρχουν για τη Μάλτα, για τη δική μου χώρα την Πορτογαλία έρευνες που βρίσκονται εν εξελίσσει. Και μάλιστα υπουργοί που, βρίσκονται στην, που βρισκόταν στην προηγούμενη κυβέρνηση της χώρας μου, αλλά και αστυνομικοί και επικεφαλής υπηρεσιών δίωξης. Αυτό δείχνει ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει άμεση πρόσβαση σε αυτές τις παράνομες ε, διαδικασίες και επιχειρήσεις και φυσικά στην ε, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Κάποιες λοιπόν από αυτές τις έρευνες ξέρω ότι έχουν ε, φτάσει και στην Eurojust και γίνονται από κοινού μεταξύ κρατών μελών και Eurojust. Όσον αφορά λοιπόν το ξέπλυμα πρόμικου χρήματος, τα γραφεία σας έχουν το απαραίτητο προσωπικό και μέσα για να μπορέσουν να δεκπεραιώσουν επιτυχώς αυτές τις έρευνες. Έχουν εντοπιστεί οι δυσκολίες και υπάρχει τρόπος να ξεπεραστούν. Όσον αφορά το Panama Papers, εμείς ξεκινήσαμε μια διερεύνηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και βεβαίως υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες στηρίζουν, αλλά κάποιες είναι μπλεγμένες σε αυτήν την ε, υπόθεση. Μπορείτε να μας πείτε πώς έχουν οι έρευνες μέχρι τώρα. Τώρα, για το PNR. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση και αξιολόγηση για το πώς προχωρούν αυτές οι έρευνες και ποιος σας στηρίζει. Εγώ βλέπω εδώ, όσον αφορά το PNR, το οποίο εξάλλου εγώ στήριξα, Και μάλιστα οι δικές μας προτάσεις συμπεριλάμβαναν στον έλεγχο και ιδιωτικά αεροσκάφη. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τους οποίους οι έλεγχοι δεν γίνονται όπως παραδείγματο χάρη ένα ιδιωτικό αεροσκάφος του, της πριγκιπικής οικογένειας Σαουδικής Αραβίας που σταμάτησε στην Ιορδανία. Ξέρουμε ότι εκεί φορτώθηκαν Ε, ναρκωτικά και ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλές τέτοιες παράνομες δραστηριότητες συνεχίζουν να ξεφεύγουν από τους ελέγχους μας. Μας πιέζει ο χρόνος αγαπητοί συνάδελφοι και βεβαίως ε, θα δοθούν αμέσως οι απαντήσεις. Έχετε πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να δώσω σύντομες απαντήσεις. Δεν ξέρω αν θα δώσω απαντήσεις σε όλους, αλλά βεβαίως μπορώ να επανέλθω και σας Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρίσμπεκ για τις ερωτήσεις σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ακούω να λέτε ότι ο συντονισμός είναι η καλύτερη απάντηση και γι' αυτό ακριβώ το λόγο θεωρούμε και εμείς ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερο συντονισμός. Θα ήθελα εξάλλου να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μας για την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίως και μας χρειάζεται αυτή η δημοσιονομική στήριξη, είναι απαραίτητη. Η απόφασή μας του 2008, το άρθρο 13 και το άρθρο 12, που προβλέπει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα συντονισμού σε εθνικό επίπεδο σε όλες τις χώρες, 28 χώρες, και βεβαίως να υπάρχει και μία ασφαλής σύνδεση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτού του Εθνικού Γραφείου και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Eurojust. Κάποιες από τις χώρες έχουν ήδη ε, αυτές τις ασφαλείς ε, επικοινωνίες το σύστημα λειτουργεί. Και βεβαίως αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, όπως ε, εξάλλου και όλα τα μεγάλα αυτά συστήματα χρειάζονται χρόνο. Πρέπει όμως εν ώψη των τρομοκρατικών επιθέσεων να επιταχύνουμε τις διαδικασίες μας Σήμερα έχουμε πολύ, πολύ καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Ευχαριστούμε όλα τα κρατημέλη που μας τροφοδοτούν με στοιχεία, με υποθέσεις. Έχουμε πολύ καλές επαφές, ενισχυμένες επαφές ε, με το Παρίσι και βεβαίως με τις κοινέ ερευνητικές μας ομάδες η ανταλλαγή πληροφών λειτουργεί με πολύ καλό τρόπο. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, προσχωρήσουν στο σύστημα αυτό. Πρέπει να έχουμε μια στάση επιμονής με μακροπρόθεσμους στόχους. Η Eurojust σαφώς και θα πρέπει να ενισχύσει την επικοινωνία της με καλύτερη επικοινωνία με ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών και το κάθε κράτος, το κάθε εθνικό γραφείο θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σύστημα ολοκληρωμένων πληροφοριών. Η Ιταλία, παραδείγματο χάρη, πολύ πρόσφατα έκανε κάποιες αλλαγές στο σύστημά της DNA και όσον αφορά την πληροφορία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συλλέγει πληροφορίες που αφορούν όχι μόνο τις δραστηριότητες της μαφίας, αλλά και ε, επιχειρήσεις που αφορούν την τρομοκρατία. Και εδώ βλέπουμε ότι οι πληροφορίες αυτές πολλές φορές διασταυρώνονται, είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Το ίδιο έκανε και η Ισπανία με την δημιουργία ενός εθνικού γραφείου μες εθνικής υπηρεσίας με εξειδικευμένο προσωπικό για να μεταβιβάζει πληροφορίες ε, εγκαίρως και με έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Βλέπουμε ότι λοιπόν τα κράτη-μέλη αυξάνουν τις προσπάθειές τους έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο μέλλον. Συμφωνία συνεργασίας, η δημιουργία ενός δικτύου και σημείων ε, συνδέσμων, επαφών όσον αφορά τις προτεραιότητές μας, την Αλβανία και την Σερβία, οι διαπραγματεύσεις ε, βρίσκονται εν εξελίξει, συνεχίζονται, συνεχίζουν οι δύο χώρες αυτές να είναι στην σειρά των προτεραιοτήτων μας πολύ ψηλά. Η προστασία των δεδομένων βεβαίως και είναι ύψιστη προτεραιότητα για την Eurojust. Και προχωρούμε πολλές φορές με μικρά ε, βήματα. Όλα αυτά λοιπόν που σας είχα πει πριν από λίγους μήνες ισχύουν. Ευχαριστώ τον Πολωνό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς δεν κάνουμε την ανάλυση των εθνικών νομοθεσιών, αλλά αυτό το οποίο κάνουμε και μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι σε όλες τις εκθέσεις μας έχουμε επιμείνει ιδιαίτερα στην ανάγκη για κοινή μεν αντιμετώπιση αλλά από την άλλη και για κοινού στόχους, δηλαδή νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες να αντικατοπτρίζουν το κοινό ψήφισμα να αντικατοπτρίζουν τις συμβάσεις ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας. Όλα αυτά είναι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται και από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής. Σε όλες τις εκθέσεις τις οποίες κάναμε μέχρι τώρα, έχουμε προσπαθήσει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τις ανάγκες. Η κοινή νομοθεσία από μόνη της δεν είναι κάτι το οποίο αρκεί. Είναι κάτι το οποίο είναι ευθύνη των κρατών μελών περισσότερο και όχι τόσο της Ευρώπης. Αλλά παρόλα αυτά και στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος και στον τομέα των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων και σε σχέση με τρίτες χώρες θα πρέπει να σεβόμεθα πλήρως το γράμμα του νόμου και στις δύο πλευρές. Έτσι θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε την ριζοσπαστικοποίηση, να βοηθήσουμε την από ριζοσπαστικοποίηση και τα προγράμματα τα αντίστοιχα αντίστοιχα με τις ε, ρυθμίσεις που ισχύουν σε επίπεδο ποινικού δικαίου σε κάθε χώρα. Να ευχαριστήσω και την επόμενη κυρία για τις ερωτήσεις της. Εγώ αναφέρθηκα στις συστάσεις και στον τομέα των χρηματοδοτικών, στον τομέα των εσόδων του, της εγκληματικής δραστηριότητας, σε στενή συνεργασία με τα δίκτυα FIU. Νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία συζητούνται όχι μόνο σε επίπεδο παράνομων δραστηριοτήτων αλλά και σε επίπεδο στρατηγικών ομάδων και για το τράφικινγκ. Γιατί τα θέματα αυτά δυστυχώς είναι επαναλαμβανόμενα αυτά τα οποία συμβαίνουν σαν παράδειγμα σε επίπεδο ψηφιακό είναι θέματα τα οποία έχουμε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία να συλλάβουμε σε εισαγωγικά, να κατανοήσουμε για να αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια. Δυστυχώς δεν μπορώ να αναφερθώ σε τρέχουσες δικαστικές διαδικασίες οι οποίες θα έρθουν στην επικαιρότητα όταν ολοκληρωθούν, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω για αυτές τώρα γιατί αυτές είναι πληροφορίες οι οποίες δεν προέρχονται από εμά, αλλά κυρίως από τα κρατη και αυτό δεν μπορώ να το αγνοήσω. Είμαστε υπέρ ε, του PNR, είμαστε ανάμεσα σε αυτούς που ζητούν την εφαρμογή του PNR, θέλουμε όμως όλα τα αποδεικτικά στοιχεία να συλλέγονται με ορθό τρόπο και να χρησιμοποιούνται με απόλυτα υπεύθυνο τρόπο και αν το σύστημα δεν είναι το κατάλληλο θα πρέπει να τροποποιηθεί. Και είμαστε στη διάθεσή, μας, στη διάθεσή σας μάλλον για περαιτέρω ανταλλαγές απόψεων. Σας ευχαριστούμε και έχουμε στείλει και αντίτυπα της αιτήσεις έκθεσης και των διαφανειών για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη. Ε, σας ευχαριστώ και περνάμε στο επόμενο θέμα, την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης. Η Επιτροπή μας, όπως ξέρετε, είναι κατ' ουσία αρμόδια για την προστασία στην επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δικαιωμάτων των πολιτών, των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων και φέρει το σημαντικό καθήκον τη εκπώνηση ετήσια έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο ψήφισμα έχει υιοθετηθεί το Σεπτέμβριο του 2015 και τώρα έχει δρομολογηθεί η επόμενη ετήσια έκθεση. Μάλιστα την περασμένη Ιούνιο είχαμε σχετική ακρόαση, οπότε που συζητήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης και πανεπιστημιακούς, τις εκθέσεις τους, πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει και τις προτάσεις τους για να διαφυλάξουμε καλύτερα τις τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ακούσουμε τώρα τον εισηγητή μας, τον κύριο Νάγκη, που θα μας κάνει την παρουσίαση της έκθεσης του. Παρακαλώ κύριε Νάγκη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. κύριε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, ε, αξιότιμοι σκιώδη ηγητές. Ε, θα ήθελα να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης με θέμα την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της έκθεση για το 2015. Ε, φυσικά αναφερόμαστε στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πολλές οδηγίες του Συμβουλίου εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευρωπαϊκές στρατηγικές και οδικούς χάρτες που λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση αυτής της έκθεσης και επίσης ε, λαμβάνουμε υπόψη και προηγούμενα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και την έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από πέρυσι. Με όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν ε, πιστεύω ότι εκπώνησα μια ισορροπημένη έκθεση που φυσικά δεν ε, έχει τη φιλοδοξία μέσα σε 13 σελίδες να καλύψει όλα τα προβλήματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και στην έκθεση του ΦΡΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ε, που είναι 60 σέλιδη, καλύπτονται περισσότερα. Εμεί έχουμε πολύ λιγότερη έκταση στι εκθέσει μα. Καλύψαμε λοιπόν πολλά θέματα τη περσινή χρονιά, αλλά και κάποια θέματα που δεν καλύπτονται συχνά από προηγούμενε εκθέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της έκθεσής μου. Φυσικά το πιο ζήτημα, μετανάστευση, ενσωμάτωση και ένταξη. Εκεί ζητούμε αποδεκτές λύσεις και κατάλληλους πόρους. Το βασικό μήνυμα είναι να τονίσουμε τη σημασία της ένταξης των μεταναστών παρά να έχουμε αναποτελεσματικές προσπάθειες ενσωμάτωσης ομάδων ε, που πολύ συχνά για τις προσπάθειες οδηγούν σε διαχωρισμό. Επίσης, ε, δεύτερο σημαντικό θέμα, ασφάλεια και καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τονίζουμε τη σημασία που έχει η σωστή αντιμετώπιση των θυμάτων της τρομοκρατίας. Σε ό,τι αφορά την εμπορία ανθρώπων, επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα στα παιδιά και στο κεφάλαιο για τα εγκλήματα μίσου, που είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα της μέρα μας, ε, λόγω της γνωστής ε, περίπτωσης ε, δολοφονίας Πολωνού ε, κατά πάσα πιθανότητα λόγω εγκλήματος μίσου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δυστυχώς δεν είχαμε αρκετές σελίδες στη διάθεσή μας για να μιλήσουμε και για τη βία κατά των γυναικών. Γι' αυτό προτιμήσαμε να αναπτύξουμε περισσότερο το θέμα των δικαιωμάτων των παιδιών ένα ζήτημα που αναφέρεται σε πολλές παραγράφους. Σε ό,τι αφορά τις μειονότητες, ε, εντοπίζουμε τα προβλήματα και καλούμε την ανάγκη ενέβρεσης ε, λύσεων στα προβλήματα των ΑΜΕΑ, των ανθρώπων με αναπηρίες, των ηλικιωμένων, των δικαιωμάτων των Ρωμά και τέλος μιλούμε για τη σημασία που έχει η συμμετοχή του πολίτη στη δημοκρατία για να δημιουργηθεί ένα θετικό αίσθημα των πολιτών για το παραδοσιακό πολιτικό βίο και για να αποκρούσουμε, να αποτρέψουμε τη βία την επιθετικότητα που είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς παρατηρούμε αρκετά το τελευταίο καιρό στην Ευρώπη. Αυτά ήταν συντομία τα βασικά στοιχεία της ε, έκθεσης μου, του σχεδίου έκθεσης. Σας προτείνω να τη διαβάσετε και περιμένω τα σχόλια και τις απορίες σας. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, η έκθεση αυτή έχει και μια προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών που λήγει στις 16 Σεπτεμβρίου. Εδώ 12 και 13 Οκτωβρίου έχουμε προγραμματίσει την εξέταση των τροπολογιών στην Επιτροπή μας. 17 Νοεμβρίου θα θέλαμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ώστε να μεταβάσουμε αυτή την έκθεση στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όντως η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 16 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νάντι. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στους Σκιώδης, ο κύριος Νίτερ Μιλέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο Γιώζεφ Νάγκη για την ε, πρόταση σχεδίου που μας έκανε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή βάση για να φτάσουμε σε μια πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση. Αναφέρει τις ε, αλλαγές από πέρσι μέχρι φέτος, από την προηγούμενη δηλαδή έκθεση και νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε πώς η κατάσταση των θημελιδών δικαιωμάτων εξελίσσεται, προοδεύει από τη μια χρονιά στην άλλη, αφού γίνεται σε αιτήσια βάση αυτή η έκθεση. Όταν συναντηθήκαμε οι σκιώδεις, εντοπίσαμε κάποιους τομείς που θα θέλαμε να δοθεί περισσότερη έμφαση στην έκθεση. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υιοθετηθεί μια τέτοια έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα χωρίς να μιλήσουμε για το κράτος δικαίου και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Έκθεσης. Στην έκθεση Ιντβέλτ αναφέρεται το θέμα αυτό ειδικότερα, αλλά νομίζω ότι η δική μας, αν θέλετε, οπτική γωνιά είναι διαφορετική και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω το θέμα αυτό. Θα ήταν σοβαρή παράληψη. Η έκθεση ΦΑΜ επίσης αναφέρεται και στα δικαιώματα των μειονοτήτων, των σεξουαλικών μειονοτήτων, της παραβιάσης των δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά και την ανάγκη να ακυρωθεί η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Το θέμα της αξιοπρέπειας των μεταναστών, της ένταξης των μεταναστών, αλλά και όλες οι διαδικασίες επιστροφής τους και επαναπρόθεσης τους πρέπει να γίνει με την ειδική αναφορά στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το ίδιο θα ήθελα να αναφερθώ και στη μειονότητα των Ρωμά, και στα τελευταία φαινόμενα εγκλημάτων μίσους αλλά και ομιλίες μίσους που γίνονται ένα σύνηθε φαινόμενο και θα αναφερθώ ειδικότερα στο τελευταίο φαινόμενο του εγκλήματος αυτού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να αναφερθούμε σε όλους τους τομείς που πρέπει να βελτιωθούν. Δεν μπορούμε να είμαστε επιλεκτικοί στην προσέγγιση μας. Βεβαίως θα προετοιμάσουμε τροπολογίες και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τις καλύτερες ε, συμβιβαστικές λύσεις και συμβιβαστικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κίπεκ από το ECR. Oh, sorry. I also, I, I also want to thank you to Mr. Και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία στην έκθεση αυτή. ασχολείται με τις πιο ευαίσθητες και ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες, τα παιδιά ιδιαίτερα. θα συμφωνήσω με τις συστάσεις αυτών οι οποίοι θέλουν να συμπεριληφθούν και οι άνθρωποι με αναπηρία. Ξέρουμε εδώ τον αγώνα που δίδει η κυρία Στίβενς, η οποία οργανώνει και μια σημαντική διάσκεψη για την πολυγλωσσία και πόσο σημαντική είναι η πολυγλωσσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τους Ρωμά. in the EU Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εδράζεται πλήρως στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, το πρώτο άρθρο έχει σχέση με την ανάγκη αντιμετώπισης με αξιοπρέπεια και νομίζω ότι το θέμα της αξιοπρέπειας είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και είναι ντροπή για τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Ξέρουμε τι γίνεται και με τα στρατόπεδα των προσφύγων, ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν και σε επίπεδο πορνείας και σε επίπεδο οργανωμένου εγκλήματος. Δυστυχώς υπάρχουν περισσότεροι σκλάβοι σήμερα από τότε που ίσχυε ε, θα έλεγα επίσημα το καθεστώς αυτό. Ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκατομμύρια άνθρωποι ε, βιάζονται, τους χορηγούν δια της βίας ε, ναρκωτικά, τους παίρνουν τα όργανα τα, του σώματός τους και παραβιάζονται συστηματικά τα δικαιώματά τους και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ντροπή. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ρατσισμού, ξενοφοβίας, ισότητας των φύλων, τραγικό θέμα για τις οικογένειες. Ε, υπάρχουν θρησκευτικές ε, διακρίσεις, ε, δογματισμοί, έλλειψη σεβασμού, αγνοώντας αυτά τα οποία έχει ζητήσει ο Ιησούς Χριστός. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση και με το άρθρο 2 των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι το πρόβλημα της, του δικαιώματος στη ζωή. Σκοτώνουμε πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες λίγο πριν ουσιαστικά τη γέννησή τους. Δημιουργούμε ένα μεγάλο δημογραφικό χειμώνα ο πολιτισμός μας στην ουσία είναι βουτυγμένος στο αίμα των αθώων παιδιών που χάνουν τη ζωή τους σε αιτήσια βάση. Ξέρω ότι το θέμα αυτό ε, κάποιοι από εσά το δέχεστε και πολλοί από εσά το απεχθάνεστε. Αλλά νομίζω ότι όσο μιλάμε παιδιά χάνουν τη ζωή τους, ε, αγέννητα φυσικά παιδιά, και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο έχουμε στη διάθεσή μας για να σταματήσουμε την κατάσταση. Να σταματήσει λοιπόν αυτή η κατάσταση και να αποδείξουμε ότι πράγματι οι αμβλώσεις δεν μπορεί να είναι τμήμα ε, της προσπάθειας για την αποκατάσταση της υγείας και της υγιεινής στην Ευρώπη. για ιατρικούς, δεοντολογικούς και δημογραφικούς λόγους θα ήθελα να σας ζητήσω να σταματήσετε την υπαριθμόν ένα παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ένωση, την άμβλωση. Ευχαριστώ. Και τώρα εκ μέρους των ελευθέρων η κυρία Μλίναρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για τη συνεργασία που είχε με τους και οδησηγητές ε, καταρτίζει ένα κατάλογο των βασικών στοιχείων σε ό,τι αφορά την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπάρχουν κάποιε παραλήψεις. Βέβαια τα σχόλιά μου ακολουθούν τελείω διαφορετική κατεύθυνση από ό,τι προλαλή σα. Εμένα με ενδιαφέρουν οι νέε προκλήσει στην ε, ελευθερία διακίνηση, στην ε, ιδιωτική σφαίρα, τη ισότητα των φύλων. Μόνο με παράγραφο αναφέρεται στη βία κατά των γυναικών και σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο για τη μετανάστευση και το άσυλο, έχω τρία σχόλια. Πρέπει να τονίσουμε καταρχήν το γεγονό ότι το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε πολλέ διαδικασίε επιβολή κυρώσεων κατά των κρατών μελών για ανεπαρκή εφαρμογή τη κοινοτική νομοθεσία, ε, ιδιαίτερα των διατάξεων για το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Επίση, ε, ο μηχανισμό επανεγκατάσταση δεν τέθηκε σε εφαρμογή στα περισσότερα κράτη-μέλη. Επίση, στην ίδια παραγραφό θα πρέπει να αναφέρουμε και το όλο και μεγαλύτερο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων και του συναφεί κινδύνου να επέσουν θύματα εμπορία ανθρώπων. Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο για την ασφάλεια, θα πρέπει και εκεί να θετήσουμε μια προσέγγιση που θα εδράζεται στα θεμελιώδη δικαιώματα και να το αναφέρουμε και στον τίτλο. Τέλος, θα ήθελα η έκθεση να αντιμετωπίζει τις αδυναμίες ε, ε, εξαιτία της ε, μη εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων από το δικαστικό σύστημα και τέλος αναφέρεται και το κράτος δικαίου. Αυτή την άκουσα θα ακολουθήσουν και οι τροπολογίες μας και προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία και με τον εισηγητή και με τους λοιπούς και εισηγητές. Ευχαριστώ. Έχουμε μήπως από την ΚΟΕ κάποιον εκπρόσωπο δεν βλέπω κάποιον από την ΚΟΕ, από τους πράσινους, σκιώδης ηγετής ή άλλος. Η FTD. Κυρία Ζίπελ. Έχω και την κυρία Γκόμες μετά στο κατάλογο. Θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη δήλωση, γιατί δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον τρόπο που μιλούμε εδώ για την άβλωση και να την εξομοιώνουμε με τη δολοφονία είναι άνω ποταμών και απαράδεκτο. Καμία γυναίκα που ποτέ δεν κάνει την άβλωση ή την έκτρωση για πλάκα ή επειδή είναι κάτι καλό. Είχαμε εκτρώσεις α, ε, α, ε, από αιώνες, ε, εδώ και αιώνες. Απλώς μερικοί ε, το θέμα είναι ή θα μπορούμε να την περιβάλλουμε κάποια χέγγια ή να την κάνουμε τρόπο που θα δημιουργεί κίνδυνο και για την έγκυο μητέρα. Απλώς ε, στις χώρες μας εδώ έχουμε πολλά παιδιά που δεν, που δεν ε, μεγαλώνουν σε αποδεκτές συνθήκες. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει πολύ περισσότερο από το ζήτημα των ογλώσεων. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη αμέριστη αποστήριξή μου προς τα σχόλια τη κύρια Ζίπελ για τι αμβλώσει. Και εγώ θα ήθελα να πω με σαφήνεια ότι με ενδιαφέρουν πολύ περισσότερα παιδιά που ήδη έχουν γεννηθεί και που ζουν σε άθλιες συνθήκε σε αφόρητη μιζέρια, παρά α, τα γέννητα παιδιά που ούτως ή άλλως και από νομική άποψη δεν είναι πρόσωπα δεν έχουν νομική υπόσταση. Επίσης, ε, νομίζω ότι θα πρέπει <clears throat> να τονίσουμε ότι η πιο καταστροφική παράβαση θεμελιωδών ελευθεριών είναι το, η εθελοτυφλία μας απέναντι στα δεινά των προσφύγων και των μεταναστών στις χώρες μας. Πολύ πρόσφατα ένας συνάδελφος στην Ελλάδα συναντήθηκε με απεγνωσμένους πρόσφυγες που δυστυχώς δεν έχουν επαναγκατασταθεί ακόμη και έχουν κολλήσει, έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα. Και συνάντησε μητέρες που ήθελαν να δώσουν σε αυτή τον Ευρωβουλευτή τα παιδιά της για να τα σώσουν. Και μάλιστα έβαλαν τα μωρά τους μερικές μητέρες στο δρόμο για να δείξουν σε τι απόγνωση βρίσκονταν. Τα άφησαν στην άσφαλτο. Και δυστυχώς εμείς κυβερνήσει μας κυρίως ε, εθελοτυφλούν σε αυτά τα δεινά των προσφύγων. Και μόνο το γεγονός ότι αδιαφορούμε για αυτούς που πριν από ένα χρόνο είπαμε ότι είναι 10.000 ε, συνόδευτοι ανήλικοι. Τώρα είναι πολύ περισσότεροι τα συνόδευτα αυτά παιδιά και ανήλικοι και έχουν γίνει θύματα στα αρπακτικά των διακινητών ή όσων θέλουν να τους χρησιμοποιήσουν για εξαγωγή οργάνων ή για τη τρομοκρατία. Αυτή είναι στοιχειώδης ε, απειλή για την απειλή και δεν το αναφέρουν. Δεν το βλέπουν οι κυβερνήσει. Θέλουμε να στηρίξουμε του πρόσφυγε, να του εντάξουμε, να του ενσωματώσουμε στην κοινωνία. Υπάρχουν και άλλου τρόπου να αντιμετωπίζουμε το μεταναστευτικό φαινόμενο, διαφορετικό από αυτό που αντιμετωπίζουμε του πρόσφυγε. Επίση υπάρχει σαφή ε, ε, ε, συνάφεια με την έξαρση των εγκλημάτων μίσους όπως αναφέρθηκε από τον συνάδελφο και το περιστατικό με τον Πολωνό και τα προβλήματα των κοινοτήτων Ρωμά σε πολλές χώρες ε, είναι μεγάλα. Βέβαια, το βασικό ζήτημα είναι το πλαίσιο του κράτου δικαίου. Και η συνάδεια που υπάρχει μεταξύ της κατάφορης παραβίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, από μεγάλες ομάδες και εντός Ευρωπαϊκής ε, και ο υποδαβλισμός της ριζοσπαστικοποίηση, η υποκίνηση της ριζοσπαστικοποίηση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να λάβει μέτρα κατά των χωρών που ε, αποδεδειγμένα πια παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα για τις θεμελιώδεις ελευθερίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η κυρία Κέγκε είναι η τελευταία εισηγήτρια. Υποστηρίζω πλήρως την συνάδελφο ζητώντας στα κείμενα να προσθεθεί και το θέμα της αυτοδιάθεσης των γυναικών. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτά που είπε η συνάδελφος πρέπει να ληφθούν υπόψη σε κάθε συζήτηση την οποία κάνουμε ξεκινώντας βέβαια από την προσπάθεια ενοχοποίησης των γυναικών όταν επιλέγουν την άμβλωση. Και πρέπει να δείξουμε τον απαιτούμενο σεβασμό προς τις γυναίκες. Θα ήθελα να προσθέσω ορισμένα στοιχεία. Στο κεφάλαιο για την καταπολέμηση του αποκλεισμού και την στήριξη των προσφύγων νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ότι στο έγγραφο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματα των μεταναστών το 2015 πρέπει να υπογραμμιστεί <clears throat> η σημασία της μετανάστευσης και η σημασία μιας αξιοπρεπούς υποδοχής για να αποφύγουμε αυτά που ζήσαμε το 2015. Το επόμενο θέμα αφορά την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι εύκολο να βάλουμε στην έκθεση αυτή ότι όπου μιλάμε για την πολιτική συμμετοχή το να αρνείται κανείς το δικαίωμα ψήφου σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο έδαφος της χώρας είναι παραβίαση των δικαιωμάτων του. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε στην αναγνώριση του δικαιώματος ψήφου των πολιτών που βρίσκονται στο ευρωπαϊκό έδαφος. Και ένα τελευταίο σημείο για την ιδιότητα του πολίτη, να συμπεριλάβουμε εδώ και την ανάγκη εναρμονισμού των διαφορετικών νομοθετικών ρυθμίσεων να αναφερθούμε σε αυτούς που γεννιούνται και μεγαλώνουν ε, στο ευρωπαϊκό έδαφος είναι αυτόματα πρέπει να θεωρηθούν Ευρωπαίοι πολίτες. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω κάποιον άλλο ο οποίος να έχει ζητήσει το λόγο. Θα δώσω ξανά το λόγο στον κύριο Νάγκη. Να σχολιάσει αυτά που ακούσαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις για τις συμπληρωματικές πληροφορίες που μας έδωσαν. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε κάποιες ε, τροπολογίες. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και καταλαβαίνω ότι πολλά θέματα δεν έχουν ενσωματωθεί καθότι δεν μπορούν να μπουν όλα σε μια τέτοια έκθεση. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν σαν κύριο θέμα κάποιους από αυτούς τους τομείς. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ενσωματώσουμε κάποια από αυτά τα θέματα στην έκθεσή μου, αλλά δεν μπορούμε να τα ενσωματώσουμε όλα, καθότι θα χάσουμε τις δυνατές προτάσεις μας ε, στους τομείς που στοχεύει η έκθεση αυτή. Τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των παιδιών. Βεβαίως όλοι θέλουμε να αναφερθούμε στο θέμα αυτό, τα θέματα της μετανάστευσης, αλλά και όλα τα άλλα θέματα που θίξατε. Συμφωνώ ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για άλλα δικαιώματα άλλων μειονοτήτων. Αλλά υπάρχουν και άλλες εκθέσεις που επεξεργάζονται τα θέματα αυτά. Συμφωνώ ότι το θέμα των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον αυτό που κάποιος είπε εδώ, το θέμα της μετεγκατάστασης των προσφύγων και της επανεγκατάστασης των προσφύγων και των υπο... το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι υπάρχουν αποφάσεις στη Γερμανία η γερμανική κυβέρνηση, οι γερμανικές αρχές ε, χρηματοδοτούν την επιστροφή κάποιων ε, προσφύγων ή κάποιων μεταναστών. Επίσης βλέπουμε την έλλειψη ενδιαφέροντος κάποιων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά αυτήν την μετεκατάσταση. Και βλέπουμε ότι βεβαίως παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ε, προσφύγων, όμως δεν είναι δυνατόν να πιέσουμε από τη στιγμή που ένα κράτος μέλος δεν θέλει, δεν επιθυμεί ε, να τους υποδεχθεί. Θα συνεχιστεί βεβαίως η συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα και τις επόμενες συνεδριάσεις που θα έχουμε και μέχρι να φτάσουμε στην Ολομέλεια βεβαίως θα συζητηθούν όλες αυτές οι πτυχές. Μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες. Περιμένουμε τις τροπολογίες σας και στην επόμενη συνάντηση στις 12 ή 13 Οκτωβρίου νομίζω ότι θα μπορέσουμε να υποβάλουμε τις ελικές ε, τροπολογίες και να τις ενσωματώσουμε. Επαναλαμβάνω και εγώ, λέει ο Πρόεδρος, ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 16 Σεπτεμβρίου. Και τώρα κυρίες και κύριοι, Είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Το επόμενο σημείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, που αφορά την Ουκρανία, θα ξεκινήσει στις 5. Έτσι έχει προγραμματιστεί. Δεν έχουμε παρόντες τους πιο σημαντικούς ομιλητές για το θέμα αυτό, υπουργό εξωτερικών της Ουκρανίας. Λυπούμε λοιπόν, αλλά θα πρέπει να διακόψουμε μέχρι τις 5. Ελάτε λίγο πιο νωρίς, λίγο πριν τις 5, μήπως είναι εδώ η κύριο μιλτέ μας και μπορέσουμε να ξεκινήσουμε λίγο πριν τις 5. Υπότιτλοι Zrazu Παρακαλώ καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει αμέσω να ξεκινήσουμε, μάλλον να συνεχίσουμε. Για τις 5.30 ακριβώς θα αρχίσουν οι ψηφοφορίες. Σημείο 5 τη ημέρης τη παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης ε, για την ε, κατάργηση των θεωρήσεων. Πρόκειται για τον κατανοησμό 539-2001 ε, που μεταφέρει και την Ουκρανία στον κατάλογο των χωρών υπηκοί των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρηση. Και στις 26 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σχετική πρόταση και τώρα η κυρία Γκάμπρι Λεπτοέλ και είναι η συγκεκριτή θα μας παρουσιάσει το σχέδιο εκθεσή τη. Και επίση να καλωσορίσω και την ε, κυρία Ολένα Ζέρκαλ, που είναι αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών για θέματα Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση στην Ουκρανία και είχε την καλοσύνη να έρθει για να ενημερώσει την Επιτροπή μα για τις εξελίξεις ε, στο διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας ε, για τις θεωρήσεις. Καλώς ήρθατε κυρία Ζερκάλ. Μην ξεχνάτε ότι στις 5.30 θα αρχίσει ψηφοφορία. Ε, οπότε σας θέλουμε παρακαλώ, παρόλο που είναι σημαντικό το θέμα, να είστε λακωνικοί και φιδωλοί στο χρόνο αγόρευσης. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Γκαμπριέλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Με ιδιαίτερη χαρά θα σας παρουσιάσω σήμερα το σχέδιο έκθεσής μου με θέμα την απελευθέρωση των θεωρήσεων για την Ουκρανία. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τις αρμόδιες Ουκρανικές Αρχές και την κοινωνία των πολιτών της Ουκρανίας αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ιδιαίτερα αγαστή συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Κατά την παρουσίαση της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είχα υποβάλει πληθώρα ερωτήσεων για την τήρηση των κριτηρίων του σχεδίου δράσης για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Και τελικά δόθηκαν ικανοποιητικέ λύσεις σε όλα τα σημεία που επισήμανα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση εντάσσεται στα πλαίσια όλο και μια στενότερη εταιρική σχέση μεταξύ Ουκρανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουκρανία είναι τέρο κλειδί τη Ευρωπαϊκής Ένωση στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονία και τη Ανατολική Εταιρική σχέση. Η συμφωνία σύνδεση που υπεγράφει τον Ιούνιο του 2014 και ταυτόχρονη κύρωση, της, κύρωση του από τη Βέρχοβνα Ράτα της Ουκρανίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2015 αποτελούν ένα χειρό μήνυμα και απόδειξη της ε, κοινή ε, επιθυμίας Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια ουσιαστική σύγκληση με βάση τις αρχές της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ολοκλήρωσης. Η άρση της υποχρέωσης ε, θεώρησης για τους Ουκρανούς πολίτες αποτελούν μια έμπρακτη απόδειξη και υλοποίηση αυτής της κοινή επιθυμίας και μία επιβεβαίωση της επιθυμίας δημοκρατικού μετασχηματισμού της χώρας αυτής και διπλά εχέγγυα ε, των υπηκών που θέλουν ε, ισοτιμία, κράτος δικαίου, μη, δια, μη διακριτική μεταχείριση και μία μόνιμη κατάργηση της υποχρέωσης ε, θεώρησης των Ουκρανών πολιτών που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, αυτή η απελευθέρωση των θεωρήσεων αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση εμβριθών και δύσκολων μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα στον τομέα τη δικαιοσύνη και των εσωτερικών υποθέσεων. Και όλα τα κριτήρια του σχεδίου δράση για θέματα ασφάλεια εγγράφων, διαχείριση ε, συνόρων και μετανάστευση, ασφάλεια ε, και δημόσια τάξη, αλλά και εξωτερικών σχέσεων και δικαιωμάτων του πολίτη, όλα αυτά τα κριτήρια έχουν ε, υλοποιηθεί. Και μάλιστα, η συγγήτρια, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στα εξή θέματα. Καταρχήν, καταπολέμηση της διαφθοράς τρεις βασικοί φορείς ε, προβλέφθηκαν για την καταπολέμηση αυτή το Εθνικό Γραφείο Πάταξης της Διαφθοράς, το Ειδικό Γραφείο για την Πρόληψη της Διαφθοράς και η Εθνική Ασφάλεια κατά της διαφθοράς. Είναι τα, οι βασικοί φορείς. Μάλιστα, τελευταία, τελευταίος αυτός ο για την πρόληψη της διαφθοράς που επικεντρώνεται στην πολιτική διαφθορά και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων θα, ε, κομμάτων θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των, των Ουκρανών πολιτών στην, ε, στην, πολιτική, ε, στην πολιτική τάξη. Και επίσης έχουμε από την 1η Σεπτεμβρίου ε, online εφαρμογή για τα έσοδα των ε, δημοσίων υπολήλων και επίσης η μεταναστευτική κίνδυνη. Θα ήθελα να τονίσω ότι το ποσοστό απόρριψης χωρίς θεώρησης ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους, ε, Ευρω... για τους Ουκρανούς είναι ελάχιστο. Είναι λιγότερο από το 2% των ε, αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. Απορρίπτονται. Επίση, η Συμφωνία Πανισδοχή Ευρωπαϊκή Ένωση Ουκρανίας για τον επαναπατρισμό των παράτυπων μεταναστών εφαρμόζεται αποτελεσματικά με ουσιαστικό ποσοστό επανεισδοχής 80%. Κάτι που αποδεικνύει την εξαιρετική συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωση Ουκρανία και μετριάζοντα τους μεταναστευτικού κινδύνου. Επίσης, ενθαρρύνω την ε, Ουκρανία να επιταχύνει την έκδοση βιομετρικών ε, διαβατηρίων και τις ε, πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα μετάβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς θεώρηση. Επίση, προσοχή να μην γίνει κατάχρηση τη απελευθέρωση των ποσοστώσεων από δίκτυα οργανωμένου εγκλήματο. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, η σύνδεση των σημείων ε, ε, των συνόρων με την βάση δεδομένων της Interpol συνεχίζεται. Βρισκόμαστε στην τελική φάση της σύναψης ε, συμφωνίας στρατηγικής και επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ Europol και Ουκρανίας. Και οι προσπάθειες που κατέβαλε η Ουκρανία στα πλαίσια του σχεδίου δράσης απελευθέρωση των θεωρήσεων θα πρέπει να συνεχίσουν να επιβεβαιωθούν ε, χρονικά, γιατί είναι σημαντικό τα κριτήρια του σχεδίου δράσης να γίνονται σεβαστά και να μην γίνει καμία παλιδρόμηση. Ιδιαίτερα σε ό,τι φορά τους φορείς ε, και τα θεσμικά όργανα που θεσπίστηκαν προκειμένου να παταχθεί διαφθορά. Και επίσης θα πρέπει να εφοδιαστούν με οικονομικούς πόρους αλλά και με την απαραίτητη πολιτική βούληση γιατί τα όργανα και τα μέσα υπάρχουν. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ να εγκρίνουν το σχέδιο έκθεση, επιβεβαιώνοντας τι αρχέ με βάση τι οποίε κάθε χώρα που πληρεί όλα τα κριτήρια ε, μπορεί να τυχεί ε, του καθεστώτου απελευθέρωση θεωρήσεων και από το σεβασμό τη μεθόδου αυτής εξαρτάται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εταίρος τρίτης χώρας, αλλά και ε, της επιβεβαίωσης ε, και της ε, επιβράβευσης μιας χώρας που ακολουθεί το, τις αρχές του κράτους δικαίου και τον σεβασμό του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ των προτέρων τους συναδέλφους για τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Γκαμπριέλ. Ποιο από του σκιώδη θα ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Για το ECR την ομάδα μας έχει μεγάλη σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβεται τους δικούς της κανόνες. στη συγκεκριμένη περίπτωση τα κριτήρια για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Πολιτικά και στρατηγικά το θέμα αυτό με την Ουκρανία έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά και πολιτικά κριτήρια. Στην τελική έκθεση προόδου η Ουκρανία έχει σημειώσει την απαιτούμενη πρόοδο και μεταρρυθμίσεις. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις και θα υποστηρίξουμε την πρόταση. Ταυτόχρονα η Ουκρανία είναι μια χώρα μεγάλη και τεράστιες οικονομικές δυσκολίες. Έχει προβλήματα επίσης διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος σε μεγάλη κλίμακα. Πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια στους τομείς αυτούς έτσι ώστε να υποστηρίξουν οι Ευρωπαίοι πολίτες την χορήγηση των θεωρήσεων. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό άρνησης χορήγησης θεωρήσεων είναι πάρα πολύ χαμηλό και το σύστημα λειτουργεί. Ευχαριστώ Γιάζεκ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι η Ουκρανία πληρεί τα απαραίτητα κριτήρια και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές είχε πάει η αντιπροσωπεία μας εκεί. Είχαμε ενδιαφέρουσες συναντήσεις με τον ε, αντιπρόεδρο, με τον πρόεδρο Ποροσένκο, με τοπικές περιφερειακές αρχές και ήμασταν σε θέση να επισκεφθούμε επίσης και ένα συνοριακό φυλάκιο ανάμεσα στην Ουκρανία και την Πολωνία και να ελέγξουμε τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές προπαρασκευάζονται για την απελευθέρωση. Από αυτά τα οποία είδαμε θα συμφωνήσουμε λοιπόν όπως και η Επιτροπή Είναι σαφές ότι οι ΜΚΟ θα θέλαμε να δούνε να γίνεται καλύτερη και γρηγορότερη προσπάθεια αντιμετώπισης της διαφθοράς. Όμως υποστηρίζουμε εν πολλής την απελευθέρωση των θεωρήσεων και πέρα από το θέμα της απλούστευσης των ταξιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η απελευθέρωση αυτή είναι και μια τεράστια ενθάρρυνση θα έλεγα προς τους πληθυσμούς έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην εγκαταλείψει χώρες όπως η Ουκρανία και να τηρήσει τις υποσχέσεις της. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Ζέρκαλ. Κατανοεί ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά έχει το λόγο. Αγαπητά μέλη, είναι με μεγάλη ικανοποίηση βρίσκομαι εδώ σήμερα και παίρνω το λόγο για την κατάσταση στη χώρα μου σε σχέση με την χορήγηση των θεωρήσεων. Το πρόγραμμα δράσης αυτό είναι ο δικός χάρτης, θα έλεγα, για τις μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία σε πολλούς τομείς που καλύπτονται. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε 144 benchmarks κεντρικούς στόχους και σε μια δεύτερη φάση 400 επιπλέον στάδια. Οι περισσότερες προϋποθέσεις έχουν πλέον εκπληρωθεί. Και εδώ εννοώ και τον τομέα καταπολέμησης της διαφθοράς τον οποίο αναφερθήκατε. Να μου επιτρέψετε να αναφέρω τα βασικά μας επιτεύγματα. Ένα από τα επιτεύγματα αυτά είναι η εισαγωγή βιομετρικών ε, διαβατηρίων. Ήδη από την εποχή του 2015 εμείς εκδίδουμε υψηλής ασφάλειας απαραβίαστα έγγραφα. 1.700.000 έχουν τυπωθεί μέχρι τώρα. Αυτό ισοδυναμεί θα έλεγα με τον αριθμό των θεωρήσεων που έχουν εκδώσει οι χώρες της Ένωσης ε, κατά τη διάρκεια της ιδίας περίοδου. Ε, για τις πλαστογραφίες από το 2007 δεν έχουν βρεθεί παραποιημένα τέτοια διαβατήρια γιατί από τότε έχουμε εξυγχρονίσει ε, το σύστημα αυτό έκδοσης ταξιδιωτικών οργάνων, διαχείρισης των μεταναστευτικών κινήσεων ε, και συλλογής των στοιχείων. Όλα αυτά επέτρεψαν θα έλεγα μια σωστή εφαρμογή, απροβλημάτιστη ε, εφαρμογή της συμφωνίας ανάμεσα στην Ένωση και την Ουκρανία. Υπάρχει δικτύωση ε, των κέντρων ελέγχου, των σημείων ελέγχου, υπάρχει σύνδεση των σημείων αυτών ελέγχου με την Ιντερπόλ και όλα αυτά θα έλεγα καθιστούν το σύστημα ικανοποιητικό. Η διαχείριση των μεθοριακών ροών βελτιώθηκε, επιτρέπει την ετήσια ανάλυση ε, του κινδύνου επιτόπου και φυσικά επιτρέπει η κατάσταση σήμερα και καλύτερη αστυνόμευση και περιπολίες στις συνοριακές περιοχές. Η συμφωνία ε, συνεργασίας με τη Eurojust υπεγράφει στις 27 Ιουνίου. Έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες και για τη στρατηγική συνεργασία με την Ευρωπόλ. Και τώρα περιμένουμε την σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το πράσινο φως του Συμβουλίου για την υπαγραφή της συμφωνίας. Η Εθνική Στρατηγική ενεκρίθη από τον πρόεδρό μας τον Αύγουστο και ο οδικός χάρτης τέθηκε σε λειτουργία το Νοέμβριο του 2015. Τα έγγραφα αυτά συνετάχθησαν σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και επιτρέπεται η παρακολούθηση από πλευράς τους της εφαρμογής τους. Καταθέσαμε τροπολογίες πρόσφατα στις νομοθετικές ρυθμίσεις για να αποφύγουμε διακρίσεις σε σχέση με, το, με φύλλο και τον γενετήσιο προσανατολισμό. Οι ε, επιθεωρήσεις που έγιναν και το 2015 και το 2016 δείχνουν ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στα συστήματα αυτά. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε τις μεταρρυθμίσεις με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς, σε συνεργασία με τις ΜΚΟ μπορέσαμε να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της ε, ευρύτατης αυτής μορφής διαφθοράς στη χώρα μας. Οι υπηρεσίες που ασχολούνται έχουν το σωστό ανθρώπινο δυναμικό πλέον και έχουν τα απαιτούμενα μέσα και είναι μια ασφάλεια θα έλεγα αυτό για την ανεξαρτησία τους και την ακαιρεότητά τους. Υπάρχουν εκατοντάδες διαδικασίες εις βάρον δικαστών, εισαγγελέων και υψηλού επίπεδου πολιτικών προσωπικότητων. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης φάσης και μέσα σε 60 μέρες, 14.000 δημόσιοι υπάλληλοι και δημοτικοί υπάλληλοι θα πρέπει να δημοσιοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης η εφαρμογή αυτή θα καλύψει πάνω από 300.000 υπαλλήλους και εκπροσώπους τοπικών αρχών, βουλευτές, εισαγγελείς, δικαστές. Δεν υπάρχει προηγούμενο στον κόσμο του μεγέθους αυτής της προσπάθειας. Ευχαριστούμε τη Μαρία Γκάμπριελ για την θετική αξιολόγηση των προσπαθειών μας και ελπίζουμε, λέει η Υπουργό Τζερκάλ, να στηρίξετε με τη θετική σας ψήφο την πορεία της χώρας μου. Και ευχαριστώ και για την δυνατότητα που μου δώσατε να λάβω τον λόγο μπροστά σας σήμερα. Σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε που ήρθατε, κύριε Υπουργέ για να λάβετε μέρος στη συζήτηση. Δεν ξέρω αν εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελε να λάβει το λόγο. Όχι. Η Σλοβακική Προεδρία ίσως. Ούτε. Άλλος κανείς. Ούτε. Ο κύριος Μπέρνι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη Μαρία Γκαμπριέλ για την έκθεσή της. Είναι σημαντικό να συγκεντρώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για να είμαστε βέβαιοι ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις, έχουν υλοποιηθεί όλα τα κριτήρια και θα καταθέσουμε και τις δικές μας τροπολογίες και θα στηρίξουμε την Ουκρανία στο δρόμο αυτό για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, γιατί αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο και για την Ουκρανική κοινωνία των πολιτών, για να αντιληφθεί ότι συνεργαζόμαστε Ουκρανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, ε, για να πάρει το μήνυμα η Ουκρανία και να επιταχύνει όλες τις μεταρρυθμίσεις για να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία. Η κυρία Γκόμες. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγητριά μας, τη Μαρία Γκαμπριέλ, για την πολύ αξιόλογη και διεξοδική της έκθεση και να συμφωνήσω με τα συμπεράσματά της. Είναι σημαντικό και για μας να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας σε έναν εταίρο που έκανε ό,τι χρειαζόταν και υλοποίηση όλες τις απαιτήσεις και από πολιτική και από στρατηγική άποψη είναι να μην αθετήσουμε τις υποσχέσεις μας προς την Ουκρανία. Ευχαριστώ την κυρία Γκάμπριελ για την έκθεσή της. Ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγητριά μας για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αφού κάνει κάποια σχόλια για αυτά που ακούσαμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν, όπως και η κυρία Υπουργός Νομίζω ότι σήμερα το μήνυμα που στέλνουμε είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για πολίτες από την Ουκρανία, μιλάμε για θεωρήσεις και βεβαίως θα παρακολουθήσουμε όλη τη διαδικασία γιατί επιτέλους πρέπει να υπάρξει αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Να ενημερώσω τα μέλη ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 15η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Θα διακόψουμε για λίγα λεπτά για να προετοιμάσουμε την ε, ψηφοφορία που θα αρχίσει ακριβώς στις 5.30. Ladies and gentlemen, could you please check... Παρακαλώ, καθίστε και ελέγξτε τι έχετε φέρει τις ε, ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας, γιατί εντός ολίγου ξεκινάμε. Right, ladies and gentlemen. Uh, λοιπόν, ξεκινάμε τις ψηφοφορίες κυρίες και κύριοι. Πρώτο θέμα, νομοθετική πρόταση που τροποποιεί τον κανονισμό 539 του 2001 που μεταφέρει και τη Γεωργία στον κατάλογο των χωρών για τις οποίες δεν ε, απαιτείται έκδοση θεώρησης για τους υπηκόους της. Κυρία Γκάμπριλη, συγκίτρια, μήπως επιθυμείτε το λόγο. Όχι, οπότε περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Τροπολογία 3 πρώτα. 3 και 4. Ψηφίζουμε μαζί τις τροπολογίες 3 και 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Αιτιολογικές αναφορές και αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1. Ε, Αιτιολογία αναφορά 3α. Ναι, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 για την αιτιολογική αναφορά 3, 3β. Ναι, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Και αιτιολογική σκέψη τροπολογία 9, άρχεται η ψηφοφορία. υπεράριθμοι στους σοσιαλιστές. Έχουμε πάρα πολλούς σοσιαλιστές στην αίθουσα. Τρομερό. Ένας υπεράριθμος παρακαλώ, ένας σοσιαλιστής σας αντισταθεί στον πειρασμό να ψηφίσει. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την έναρξη των διαπραγματεύσεων και τη σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στο δεύτερο θέμα με το οποίο θα ψηφίσουμε το σημείο 7 Κυρία Χολμάιερ Θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση για το μέρος του ΕΛΚ για την ψηφοφορία. Λυπόμαστε λοιπόν, πάρα πολύ που δεν μπορέσαμε να περιμένουμε μέχρι να έχουν τηρηθεί όλα τα κριτήρια για το Κόσοβο. Γιατί ακριβώς αυτό απαιτήσαμε από άλλους και δεν το κάνουμε εδώ με το Κόσοβο και αυτή τη στιγμή γίνεται η ψηφοφορία και θα ήθελα να ληφθεί υπόψη αυτό που λέω. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί δεν τηρούνται τα ίδια κριτήρια και τα ίδια πρότυπα εδώ για το Κόσοβο. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι υπάρχουν <clears throat> δύο μέτρα και δύο σταθμά. Λυπούμε πάρα πολύ. Και όταν μιλάμε βεβαίως για απελευθέρωση θεωρήσεων με χώρες όπως την Τουρκία, θα πρέπει να τηρούμε ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές όπως και με άλλες περιοχές. Λυπούμε λοιπόν πάρα πολύ που σήμερα ψηφίζουμε για το θέμα αυτό και βεβαίως ε, το ΕΛΚ ε, θα ήθελε αυτή την θέση και αυτή την τοποθέτηση να τη λάβετε υπόψη σας. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Σύμφωνα με τους κανόνες που τηρούμε, που θα έπρεπε να τηρούμε, εάν υπάρχουν αντιρρήσεις όσον αφορά την ημερήσια διάταξη. Αυτό θα πρέπει να γίνεται εγκαίρος και όσον αφορά τη συζήτηση για την ημερήσια διάταξη. Κανείς όμως δεν έχει εκφράσει για αυτήν την ημερήσια διάταξη και για αυτή την ψηφοφορία καμία παρατήρηση και κανένα σχόλιο. Λυπούμε, αλλά εάν δεν συμφωνούν όλοι οι υπόλοιποι, θα πρέπει να τηρήσουμε την ημερήσια διάταξη και να προχωρήσουμε όπως έχει αποφασιστεί. Κυρία Χολμαϊρ, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που θέλει να πάρει το λόγο και να πει κάτι σε σχέση με αυτό που, που είπατε, που έχει αντίθετη άποψη από εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ χαίρομαι γιατί αναφερθήκατε στις αλλαγές της ημερήσιας διάταξης, κάτι που πρέπει να γίνεται εγκαίρος. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες γι' αυτό. <laughs> και αυτό γίνεται στην αρχή της συνεδρίασης κάθε φορά. Αναρωτιέμαι λοιπόν, τι έγινε από τις 3 σήμερα μέχρι τις 5.30 ξαφνικά είναι απαραίτητο να βγει αυτό το θέμα από την ημερήσια διάταξη. Ποιο είναι ο λόγο. Θα ήθελα επίση να σχολιάσω και κάτι άλλο. Βεβαίω η απελευθέρωση των θεωρήσεων δεν μπορεί να ξεκινήσει και να γίνει πριν τηρηθούν όλα τα κριτήρια. Και εννοείται ότι μόνο και εφόσον όλες αυτές οι προϋποθέσεις και οι όροι τηρούνται, θα μπει στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας αυτό το θέμα. Σήμερα όμως νομίζω ότι μπορούμε εδώ να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Να πω κάτι στον επικεφαλής της Επιτροπής. Ανακοίνωσα στον πρόεδρο της Επιτροπής την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι πρώτη φορά λοιπόν που κάνω αυτή την δήλωση. Καταλαβαίνετε όμως ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάστασή μου. Εγώ εδώ ουσιαστικά έχω μία ημερήσια διάταξη και κάθε φορά δίνω τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε έχει κάποια αντίρρηση με ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης να το συζητήσουμε. Αυτό γίνεται πριν υιοθετηθεί επισήμω η ημερήσια διάταξη. Και αυτό έγινε και σήμερα. Από τη στιγμή όμως που έχει υιοθετηθεί η ημερήσια διάταξη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την τροποποιήσουμε. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Λυπούμε όμως, αλλά πρέπει να πάρω μια απόφαση. Η απόφαση δική μου βεβαίως Μπορεί να σας φανεί δύσκολο να ανατραπεί μετά από εβδομάδες. Σε πάση περιπτώσει όμως, δυστυχώς αυτή τη στιγμή πρέπει να τηρήσουμε την ημέρα διάταξη και πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Παίρνω λοιπόν αυτή την απόφαση και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία και η τελευταία εξάλλου ψηφοφορία της ημέρας. Πρόκειται για το 539 του 2001 για την ε, ενσωμάτωση του κοσυφοπεδίου στις χώρες που, δεν, που απαλλάσσονται από θεωρήσεις, η κυρία Φαγιάννη. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ψηφοφορία, διότι στέλνουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό μήνυμα προς την χώρα αυτή, ότι είμαστε σοβαροί και ότι καλούμε το Κόσοβο να κάνει τις τελευταίες προσπάθειες έτσι ώστε να τηρήσει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια έτσι ώστε να του δοθεί το πράσινο φως για την ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα Όλες οι προϋποθέσεις υπάρχουν για να ψηφίσουμε και ζητώ από όλους τους ε, συναδέλφους ε, να στήριξουν ε, τις θέσεις μας αυτή την ψηφοφορία. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Τροπολογίες 1 και 2, οι οποίες είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Πάλι έχουμε πρόβλημα με τους σοσιαλιστές. Υπάρχει ένας επιπλέον. Σας παρακαλώ πολύ, μην δημιουργείτε δυσκολίες. Είσαστε εντάξει τώρα με τους αριθμούς. Ναι, τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία αυτή. Και τώρα περνάμε Παράγραφο 1, άρθρο 1, εισαγωγικά, τροπολογία 10. Τροπολογία 10 ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Όχι. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Απορρίπτεται. Άρθρο 1, παράγραφος 1, παράδειγμα 2, 4. Πρόκειται για την τροπολογία 11, αρχή της ψηφοφορίας, τροπολογία 11. Τέλος. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην αιτιολογική αναφορά Τροπολογία 1-3. Τέλος. Απορρίπτεται. Ετολογική σκέψη 2, τροπολογία 4. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Αιτιολογική αναφορά 4, τροπολογία 5. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. Ιτολογική σκέψη 3, τροπολογία 7. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Για το ξεκίνημα των ε, διαπραγματεύσεων και την σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Αυτό απορρίπτεται. Χρειαζόμαστε την απόλυτη πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Τέλος της ψηφοφορίας, τέλος συνεδρίασης. Just before you leave, uh, any other business? Υπάρχει κάτι για τα διάφορα. Δεν έχω σημειωμένο τίποτα στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 3 το απόγευμα εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά και στις 12 Σεπτεμβρίου, στις 7 έως τις 10 θα συναντηθούμε στο Στρασβούργο στην ειδική μας συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος της συνεδρίασης.